Αγαπητοί φίλοι, ξαναξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Τελειώσαμε τη συνεδρίαση των συντονιστών και ε, θα χρειαστεί να περιοριστείτε στη δικιά μου προεδρία διότι όλοι οι υπόλοιποι ξεφύγανε και έτσι θα συμπάσχουμε σήμερα. Οπότε ξεκινώ και σας ανακοινώνω ότι θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας με το θέμα 11 που είναι η χρηματοδότηση της αλλαγής της, του κλίματος αρχή της προσθετικότητος. Οπότε θα παρουσιαστεί μία μελέτη σχετικά με τη συμπλήρωση ε, της χρηματοδότησης η οποία ε, είχε ε, συμπληρώσει την πρόταση του DCI διότι θα πρέπει να δούμε εάν το θέμα αυτό πρέπει να προσθεθεί το 0,5 7% ε, που είναι ο στόχος διότι ε, εφόσον πρόκειται για μία δραστηριότητα η οποία απευθύνεται στην ανάπτυξη πρέπει να συνάδει με την ε, αναπτυξιακή βοήθεια στα πλαίσια αυτά πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση της ε, κλιματικής αλλαγής ε, δεν θα απορροφήσει την ε, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτήσεως που θα έπρεπε να αφιερωθεί σε άλλους στόχους αναπτυξιακούς όπως η παιδεία και η ε, υγεία. Ε, θέλω να καλωσορίσω εδώ την κυρία Ιρέν Κνόκε, ερευνήτρια στο Γερμανικό Ινστιτούτο Βίντ, η οποία προσπάθησε να διευκρινίσει το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μας με τόσο μικρή προειδοποίηση και θα έχετε επαρκή χρόνο για να μας αναπτύξετε το θέμα σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω εδώ αυτή τη μελέτη. Επειδή δεν έχω και τόσο πολύ χρόνο θα περάσω στα γρήγορα τις πρώτες διαφάνειες διότι οι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε το πλαίσιο. Η συμφωνία της Κοπενχαϊκής και η συμφωνία του Κανκούν έχει αποδείξει ότι το 2012 έχουμε 30 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία διετέθησαν από το 2010 ως το 2012 αλλά πρέπει να αυξηθεί το ποσό αυτό και από το 2020 προβλέπουμε Βλέπετε ότι το χρόνο θα διατίθενται 100 δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση υπο ε, ε, υποανάπτυξη χωρών. Είναι νέα θέματα αυτά, δηλαδή προστίθενται στην προηγούμενη χρηματοδότηση του κλίματος και επιπλέον ε, θα προσθεθούν στους, στην υπάρχουσα χρηματοδότηση για τους στόχους ανάπτυξης και επιπλέον η ε, ε, η χρηματοδότηση του κλίματος ε, έχει περιοριστεί. Πέραν αυτού θα προέρθει από πολλές πηγές εθνικές, πολυεθνικές, ε, μονομερείς, πολυμερείς, ε, μεγάλη ποικιλία πηγών χρηματοδότησης ε, για να μπορέσει να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων. Πέραν αυτού υποθέτω ότι γνωρίζετε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της ανάπτυξης και ότι είμαστε μακριά από το στόχο του 0,7% αλλά προφανώς ο στόχος αυτός δεν είναι πεπερασμένος και μάλλον το αντίθετο. Δηλαδή η κλιματολογική αλλαγή είναι ένα θέμα που προκαλεί άλλα επιτεύγματα και γι' αυτό πιστεύω ότι οποιοδήποτε ορισμός θα πρέπει ε, να προσπαθήσει να μην αποκλίνει από το στόχο του 0,7%. Οι ανάγκες διαφέρουν πάρα πολύ όπως θα δείτε από τους αριθμούς που παρατίθενται και αυτοί δεν είναι δικοί μου υπολογισμοί αλλά της Παγκοσμίας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως άρα αξιόπιστη και όπως βλέπετε ε, το, ε, τα 100 δισεκατομμύρια ε, δολαρίων είναι μάλλον ανεπαρκής για να υπάρξει και κάλυψη των αναγκών και προσαρμογή. Γι' αυτό και μιλάμε για προσθετικότητα και για τις πηγές από τις οποίες πρέπει να προέρθει αυτή η χρηματοδότηση. Επιπλέον, όπως είπα και προηγουμένως η κλιματική αλλαγή θέτει σε κίνδυνο ε, τις, ε, τις, τους στόχους που έχουμε θέσει και αναφέρεται ε, και της, ε, ε, τις ε, διάφορες τους διάφορους τρόπους να αποφύγουμε την ευαισθησία θα πρέπει να υπάρξουν γεωγραφικές προτεραιότητες και όλα τα θέματα είναι στενά συνδεδεμένα θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα προσαρμογής και βλέπετε εδώ ότι έχουμε μεγάλες γεωγραφικές προτεραιότητες παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι πολλές στοχές χώρες οι οποίοι είναι αναπτυξιακοί ε, εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι πολύ ευάλωτοι λόγω των κλιματολογικών αλλαγών όπως άλλωστε και τομείς οι οποίοι έχουν σχέση με την διατροφική ασφάλεια ή την μείωση της φτώχειας. Ε, γι' αυτό και η ύπεθρος είναι ένας τομέας ο οποίος αναφέρεται σε αυτές τις δραστηριότητες της προσαρμογής στις κλιματολογικές αλλαγές. Πέραν αυτού όμως οι δραστηριότητες σχετικά με τις κλιματολογικές αλλαγές δεν θα είναι αυτές που θα επηρεάσουν ριζικά τη μείωση της φτώχειας και είδαμε ότι μπορούν να υπάρξουν αλλαγές ε, και εάν μόνο χρηματοδοτήσει κανείς βάση των ε, αναγκών προσαρμογής δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τις προτεραιότητες τόσο γεωγραφικές όσο και τομεακές γι' αυτό και χρειάζεται η αρχή αυτή της προσθετικότητος. Θα πρέπει να υπάρχουν συνέργειες, παραδείγματος χάρη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και ενεργειακές πηγές θα πρέπει να τονίσουμε ότι στις μεγάλες οικονομίες θα χρειαστεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση διότι αυτές ρηπαίνουν περισσότερο ή μάλλον συμβάλλουν πολύ περισσότερο στις εκπομπές και ε, αυτό μπορεί να αποκλίνει από τις φτωχότερες, να απομακρύνει από τις φτωχότερες χώρες την αναγκαία χρηματοδότηση ε, και θα δούμε άλλωστε ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να ε, αποδώσουν μετά από σειρά ετών και θα χρειαστεί μεταξύ κάποιο αντισταθμιστικό μέτρο η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων μεταξύ κλίματος και αναπτύξεως είναι θέμα αποτελεσματικότητος και γι' αυτό θα χρειαστεί ε, ε, σημαντική χρηματοδότηση ακριβώς διότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Στη μελέτη προσπάθησα να επεξεργαστώ και διάφορες εναλλαστικές λύσεις, δηλαδή πόσο θα καθορίσουμε την προσθετικότητα για να τη μετρήσουμε χρειαζόμαστε μία βάση από την οποία θα ξεκινήσει αυτή η προσθετικότητα μπορούμε είτε να πάρουμε το στόχο του 0,7% που προανέφερα δηλαδή 0,7% ε, συν οποιοδήποτε ποσό. Και αυτό είναι ε, πιο, πιο συνεκτικό διότι αυτή είναι μία δέσμευση η οποία έχει ληφθεί από καιρού. Άλλη δυνατότητα είναι να πάρουμε το τωρινό επίπεδο της χρηματοδότησης για το κλίμα ε, και παραδείγματο χάρη να πάρουμε το επίπεδο του 2009 πριν από τη Συμφωνία της Κοπεχάγης. Δηλαδή οποιαδήποτε χρηματοδότηση ε, θα πρέπει εφόσον ε, ξεπερνά το επίπεδο του 2009 να είναι επιπρόσθετη και αυτό τεχνικά είναι εφικτό και μπορεί να μετρηθεί και για τις χώρες του ΩΣΑ και για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι στο σύστημα των πιστώσεων αναφέρονται προς τον ΩΣΑ αυτά τα στοιχεία αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ότι ε, εφόσον το αναπτυξιακό ταμείο είναι ήδη υψηλό, θα χρειαστεί ενδεχομένως αντί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός να υπάρχει ανακατάταξη των πιστώσεων. Στη Γερμανία παραδείγματος χάρη βλέπετε ότι ελάχιστη χρηματοδότηση για τις κλιματολογικές αλλαγές μπορεί ε, όντως να θεωρηθεί ότι είναι μία πρόσθεση σε αυτήν που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη λύση θα ήταν να θέσουμε ένα έτος αναφοράς που είναι όταν οι δότες ξεκίνησαν να χρηματοδοτούν αλλά τότε δέχεται εάν πάρουμε κάποιο χρόνο μακριά πίσω να είναι ένα μειονέκτημα. Ε, επίσης, ε, αν δεν υπάρχει μία ε, σταθερή βάση θα μπορέσουμε να πάρουμε την τρίτη εναλλακτική λύση η οποία όμως μπορεί να ισχύσει μόνο εάν είναι προσθετική δηλαδή θα μπορεί κανείς να διπλομετρήσει κάτι να υπολογίσετε ε, χρηματοδότηση του κλίματος σαν χρηματοδότηση για τη βελτίωση του κλίματος και αναπτυξιακή βοήθεια αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει στην περίπτωση αυτή ότι το ποσό αυξάνεται πέραν της χρηματοδοτήσεως της κλιματικής ε, ε, αλλαγής. Επίσης ε, θα επανέλθω αργότερα σε ένα άλλο θέμα που είναι οι χρονικοί περιορισμοί, δηλαδή μέχρι πότε θα μπορούν να ισχύσουν αυτές οι διπλές μετρήσεις. Βέβαια, εάν αναφερθούμε μόνο στις νέες πηγές δεν θα υπάρξει διπλή μέτρηση και δεν ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι στο παρελθόν υπήρχε χρηματοδότηση για την κάλυψη των ε, κλιματικών στόχων αλλά τα ποσά αυτά ε, θα είναι πολύ χαμηλά ιδίως για χώρες οι οποίες δεν φτάνουν καν στο στόχο του 0,7% και τέλος Ε, αντί κανείς να εξετάσει ε, πού καταλήγει η χρηματοδότηση θα μπορούσε να κατατάξει τη χρηματοδότηση αναλόγως των πηγών, δηλαδή από πού προέρχεται. Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα κριτήρια που προανέφερα και τεχνικά και πολιτικές σκοπιμότητες θα πρέπει να καταταξει τη χρηματοδοτηση αναλογως των πηγων δηλαδη απο που προερχεται επισης πρεπει να λαβετε υποψη σας ολα τα κριτηρια που προανεφερα και τεχνικες και πολιτικες σκοπιμοτητες θα πρεπει να συνυπολογιστουν και βλέπετε εδώ στον πίνακα αυτό ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση η οποία να επιτυγχάνει και να καλύπτει όλα τα κριτήρια. Βέβαια η πρώτη εναλλακτική λύση η οποία ε, έχει μεγάλη εφαρμοστικότητα, δεν έχει πολιτική κάλυψη ε, και για μένα η καλύτερη λύση είναι η δεύτερη και οποιοδήποτε ορισμός θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Φτάνοντας όμως το κρίσιμο σημείο τώρα, δηλαδή την πολιτική αποδοχή, βλέπετε ότι το πλέον αποτελεσματικό στοιχείο είναι το δεύτερο το οποίο όμως μπορεί να οδηγήσει σε ε, μία παρέκκληση των ε, στόχων της χρηματοδότησης και ε, γι' αυτό βλέπετε ότι θα επανέλθω στον πίνακα αυτό και ε, να σχολιάσω τις ε, τις επιλογές 1 και 3 για να σας πείσω ότι η επιλογή νούμερο 1 είναι πολιτικά πιο, μπορεί να γίνει πολιτικά πιο αποδεκτή. Τέλος βλέπουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να καταλήξει σε έναν κοινό ορισμό μέχρι το 2013 και ζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να ε, καθορίσουν την χρηματοδότηση για το κλίμα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο στόχος και βλέπετε ότι ε, είναι πολύ διαφοροποιημένος διότι υπάρχουν ε, διάφοροι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται δηλαδή έχουμε τις χώρες οι οποίες βρίσκονται εις ε, το μπλε ε, επίπεδο ε, και εδώ βλέπετε ότι εις τα κράτη-μέλη αναφέρεται το έτος αναφοράς, δηλαδή τα περισσότερα κράτη χρησιμοποιούν σαν έτος αναφοράς το 2009 ή το 2010 και όσον αφορά τη σειρά των τομέων που ε, ε, κατάταξη των χρηματοδοτήσεων είναι στο υπαριθμό 3 αλλά στο κόκκινο, στο κόκκινο τμήμα βλέπετε ότι εκεί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στη χρηματοδότηση και υπάρχει ε, μία χρηματοδότησης η οποία ε, εάν αποδοθεί περισσότερο στους κλιματικούς στόχους ε, μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί περισσότερο για άλλες σκοπιμότητες. Τέλος βλέπουμε ότι κάθε χώρα θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει το δικό της ποσοστό αλλά ε, τελικά ο στόχος μας είναι τουλάχιστον το 0,7% και ξέρετε ποιες είναι οι ε, τέσσερις χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται εδώ, αυτές που έχουν ήδη επιτύχει το 0,7%. Ε, υπάρχουν βέβαια και άλλες δυνατότητες για άλλους ορισμούς, αλλά υπάρχουν 8 χώρες που θα μπορούσαν να περιληφθούν εις το ο κόκκινο τμήμα αλλά ενδεχομένως μπορείτε να έχετε ένα πιο λεπτομερή ε, ορισμό ε, με τα στοιχεία τα οποία έχω παραθέσει εδώ. Πώς θα επιτευχθεί η προσθετικότητα. Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να μην υπάρχει παρέκκληση, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μία κατάταξη της σειράς προτεραιότητας χρηματοδοτήσεως από την οποία δεν θα αποκλίνει κανείς και θα είναι υποχρεωτική για να μην ε, ε, παρεκκλίνει η χρηματοδότηση από τους στόχους του κλίματος και να αποδίδεται αλλού και θα χρειάζεται να παρακολουθείτε ε, περισσότερο διότι είναι ένα πιο βασικό θέμα από ότι ο στόχος του 0,7%. Τέλος, η διαδρομή προς την επίτευξη του στόχου του 0,7% προβλέπει ότι θα χρειαστεί να αυξήσουμε την πολιτική αποδοχή, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν επιτευχθεί να διπλοϋπολογίσουμε και εάν δείτε το, την ισχύουσα κατάσταση σαν σημείο κινήσεως αυτό σημαίνει ότι ε, για το έτος 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και οι χώρες DAC έχουν ε, προβλέψει ότι θα πάει το μεγαλύτερο ποσοστό στην κάλυψη των ατελειών και το μικρότερο ποσοστό μόνο το 20% στην ε, την επίτευξη νέων κλιματικών στόχων. και θα προσπαθήσουμε να μείνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στο ε, πρόγραμμα δράσης ε, με τα 12 σημεία να φτάσουμε δηλαδή ε, την βοήθεια αυτή στο 0,7 ε, του GNI. Έτσι λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να σημειωθούν για θέματα ανάπτυξης να αυξηθούν κατά 0,7%, να φτάσουν μάλλον το 0,7% το 2015. Βέβαια υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις ανάμεσα στην αναπτυξιακή βοήθεια και στη βοήθεια προσαρμογής. Και γι' αυτό νομίζω ότι ούτε οι στόχοι ας πούμε για την αντιμετώπιση των λογικών αλλαγών δεν θα πρέπει να περάσουν το, 7, το 0,7%. και εφόσον όλα τα συμπεριλάβουμε και τις δύο αυτές μορφές, τους δύο αυτούς στόχους χρηματοδότησης, θα φτάσουμε το 2020 το αργότερο σε κάτι πάνω από 0,7%. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος Γκέρενς γιατί εδώ κάτι δεν καταλαβαίνω. Είπατε ότι το 2010 το 12% των ποσών δόθηκαν για την καταπολέμηση των συνεπειών και 12% για προσαρμογή. Αυτό είναι 20, είναι 24%. Όχι λέει η ομιλήτρια, 7%. Είπα 7% για την προσαρμογή και 12% για την αντιμετώπιση των συνεπειών, την μετρίαση των αρνητικών συνεπειών. Θα πρέπει νομίζω να ισορροπήσουμε τα δύο αυτά ποσοστά και ε, προσθέτοντας το 0,7% ε, στο άλλο 0,7% να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική ισορροπία. Αυτό το ποσοστό θα πρέπει να μειωθεί λοιπόν σταδιακά έτσι ώστε το 0,7% στόχος συν. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει επιλογή παρίθμου 1. Ένας ορισμός δηλαδή ο οποίος ε, θα γίνει πλήρως ε, εφαρμόσιμος ε, το 2020 το αργότερο. Ένα ακαθόδες θέμα είναι το από πού θα έλθουν τα, οι πιστώσεις αυτές, τα χρήματα αυτά. Είπαμε ότι απαιτείται να υπάρχει μια ποικιλία πηγών χρηματοδοτήσεων, δημοσίων, ιδιωτικών, πολυμερών, μονομερών, όλα έχουν εξεταστεί έτσι ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα α, χρηματοδότησης. Ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά είναι εφικτά αλλά και πάρα πολύ δύσκολο να τα πετύχουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στα χρήματα τα οποία έχουμε πει, δηλαδή 100 δις. Όλα είναι εφικτά αυτά μέχρι το 2020, αλλά να μην ξεχνάμε όμως και τις συζητήσεις ε, για τις καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τη χρηματοδότηση για την μετρία των επιπτώσεων των χρηματολογικών αλλαγών. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εδώ να δούμε τι θα γίνει με τη χρήση του φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές όταν εφαρμοστεί και πώς μπορεί ο κλάδος αυτός των χρηματοδοτήσεων να πάρει χρήματα και από εκεί. Σε πολλές ε, χώρες ε, υπάρχει λοιπόν η αρχή μέσω των εσόδων των φορολογικών να πηγαίνουν ε, στον προϋπολογισμό και από εκεί να αδιαιρούνται και να οδεύουν προς συγκεκριμένους τομείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή θα λέγαμε εκ των προτέρων σημείωσης ενός φόρου για ένα συγκεκριμένο στόχο. Αλλά παρόλα αυτά Υπάρχει δυνατότητα χρήσης φόρων για οικολογικούς λόγους, περιβαλλοντικούς λόγους και υπάρχει η δυνατότητα ένα μεγάλο ε, ποσοστό θα έλεγα των νέων φορολογικών εσόδων να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους τους οποίους ανέφερα για το 0 αυτό 7% κάτι το οποίο μπορεί και τελικά να ελαφρύνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς άλλες πηγές υψηλών δυνατοτήτων που έχουν ε, εντοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα σταθεροποιημένο σύστημα συναλλαγών για, από το εκπομπές ε, καυσαερίου. Έχει αναλάβει βέβαια μια υποχρέωση μείωσης ε, κατά 30% και όχι 20% εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θα σταθεροποιήσει τις τιμές. Η στοχοθέτηση θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη να μην μείνουμε στο 50% το οποίο αναφέρεται, στο 15% το οποίο αναφέρεται, των εσόδων δηλαδή των φορολογικών να προορίζονται για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών χρηματοδοτήσεων, να καλύπτουν τέτοιου είδους ποσοστά. Αυτό το επίπεδο τουλάχιστον κατά 25% δηλαδή θα πρέπει να καθοριστεί τώρα και να αυξηθεί ίσως και στο μέλλον, γιατί όχι. Ε, υπάρχουν βέβαια και άλλες δυνατότητες φορολογικών πηγών εδώ. Ο φόρος σαν παράδειγμα για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές είναι μια πηγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σωστά, σωστότερα από ό,τι γίνεται σήμερα το θέμα του φόρου που προέρχεται από την εμπορία των εκπομπών καυσαερίων. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό που ονομάζουμε σήμερα αρνητικές συμπεριφορές ή κακές συμπεριφορές. Τώρα πώς θα δίδονται τα χρήματα. Έχει μεγάλη σημασία οι προτάσεις του MFF και του DCI να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχουν οι δραστηριότητες για τις κλιματολογικές αλλαγές. Το DCI πρέπει να αυξήσει τα μέσα του. Έχει ένα θεματικό μέσο. Υπάρχουν επίσης σημαντικά επιπλέον κλιματολογικά μέσα και λέγεται ότι το 50% το οποίο αφορά τα αγαθά τα οποία γίνονται αντικείμενο εμπορίου και δεν ξεπερνάει το 25% του συνολικού ποσού. Επίσης το ίδιο το mainstreaming θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα επιμέρους γεωγραφικά προγράμματα και από εκεί μπορεί να υπάρξει μια μικρή αύξηση. Όλα αυτά είναι θα έλεγα καλές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των προγραμμάτων ελέγχου των κλιματολογικών συνεπειών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εκκρεμότητες. Καταρχάς τα ποσά, οι πιστώσεις αυξήνονται περισσότερο φυσικά οι ανάγκες πιστώσεων από ότι οι προϋπολογισμού του DCI. Οπότε δεν φτάνουμε στα επίπεδα τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει, το λεγόμενο benchmark. Αν δείτε τις προτάσεις για τον DCI θα καταλάβετε ότι δεν καλύπτουμε το σύνολο των αναγκών. η αρχή της μη διάχυσης αν θέλετε, απόκλησης μάλλον, είναι κάτι το οποίο άπτεται με την σωστή εφαρμογή των θυματολογικών προγραμμάτων ένα παράδειγμα εδώ, θέματα φύλου. Είναι θέματα που έχουν κάποια σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές ή όταν μιλάμε για τη δημοκρατία και δημοκρατικές εξελίξεις σε διάφορες χώρες. Είναι θέματα τα οποία άπτονται με των κλιματολογικών αλλαγών αλλά αγνοούμε συνήθως. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν καθορίζονται σωστά στον DCI έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την προσθετικότητα με σωστό τρόπο. Μία κατευθυντήρια γραμμή θα είναι σαν παράδειγμα η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των σχετικών με το κλίμα στο εσωτερικό του DCI να μην αυξηθεί ποσοστιαία περισσότερο από το ποσοστό αύξησης του συνόλου των οικονομικών δυνατοτήτων του DCI. Και τέλος, η χρηματοδότηση προς το DCI θα συγκεντρώνεται κυρίως στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Οπότε τα θέματα που αφορούν τα φύλλα στα γεωγραφικά μέρους μέσα θα πρέπει να έχουν σαν στόχο περισσότερο την προσαρμογή και όχι τόσο την αντιμετώπιση των συνεπειών. δηλαδή ε, χρηματοδότηση ε, από τη μία της προσαρμογής και χρηματοδότηση από την άλλη της αντιμετώπισης των επιπτώσεων θα πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Για τις συστάσεις τώρα, κλείνοντας αυτά τα οποία σας προείπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσει και να προωθήσει με ένα κοινό ορισμό της προσθετικότητας, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί εδώ. Σύμφωνα με την σημερινή πρακτική αναφορά της δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, αυτό θα θέσει σε μειονεκτική προσωρινά θέση τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ένας κοινό ορισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι αρκετά πιο φιλόδοξος από ότι οι ορισμοί τους οποίους χρησιμοποιούν άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη μια τέτοια κίνηση θα, θεωρη, ειδωθεί ευνοϊκά από τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια γιατί διασφαλίζεται ε, υψηλό επίπεδο διαφάνειας, δυνατότητα προγραμματισμού και αυτό θα πιέσει και τις άλλες χώρες να συμφωνήσουν στα δικά μας επίπεδα γιατί όλοι συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρωτοπόρο στον καθορισμό των μέσων τα οποία είναι χρήσιμα. Κάθε ορισμός θα πρέπει να μένει επίσης, να εμένει θα έλεγα στο πρόγραμμα αυτό των 12 σημείων και στο 0,7% το οποίο ίσως θα πρέπει βέβαια να αναθεωρηθεί στο μέλλον γιατί οι ενδιάμεσοι στόχοι δυστυχώς δεν έχουν επιτευχθεί σε πάρα πολλές ε, χώρες. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, Κάθε ορισμός θα πρέπει να εμείνει στο 0,7% και να επιτρέψει τη διπλή συμπερίληψη. Και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα τώρα, θα πρέπει να καταλήξουμε σύντομα σε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη του 0,7% συν. 0,7 συν. Και αυτό το 2020. Είναι προϋπόθεση για την διπλή συμπερίληψη αυτό. Να αναπτυχθούν και να αυξηθούν όλα τα επίπεδα. για τις υπόλοιπες συστάσεις τώρα σχετικά με το MFF και το DCI. Νομίζω ότι εδώ είναι απλά τα πράγματα. Είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτά, αλλά το MFF θα πρέπει να δώσει περισσότερες πιστώσεις για τις κλιματολογικές αλλαγές. Απαιτούνται περισσότερες πιστώσεις, γιατί έχω ένα διπλό καπέλο εδώ. Είναι, ξέρω, δύσκολο στον τομέα των, της, της αντιμετώπισης των κλιματολογικών συνεπειών να βρει κανείς πηγές κλιματοδότησης. Από την άλλη όμως, αυτή η βοήθεια όταν ευρεθεί δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των αναπτυξιακών στόχων. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η προσθετικότητα, πρέπει να δοθούν εγγυήσει για την προσθετικότητα σε σχέση με τις αναπτυξιακές ισχύουσες δραστηριότητες και στόχους. Και όπως έχω ήδη πει, η ισορροπία ανάμεσα στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στην προσαρμογή θα πρέπει να καθοριστεί με σωστό τρόπο και να εμείνουμε περισσότερο στην προσαρμογή. Στο μέλλον το 2 τρίτα θα πρέπει να πηγαίνουν στην προσαρμογή. Το DCI συγκεντρώνουν την προσοχή τους στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και έτσι η προσαρμογή για τις χώρες αυτές είναι μάλλον πιο σημαντική από την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών. Και τέλος, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις χώρες της λεγόμενης μεσαίου εισοδήματος γιατί σβήνουν λίγο από τον DCI σιγά σιγά και χρειάζονται ίσως ένα διαφορετικό μέσο το οποίο να καλύπτει τις δικές τους ανάγκες. Είναι χώρες μεσαίου εισοδήματος οι οποίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν ανάγκη από δημόσιους χρηματοδοτήσεις και για προσαρμογή και, αντιμετώπιση των, και για αντιμετώπιση των συνεπειών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση περισσότερο με τον DCI αλλά περισσότερο με το MFF. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κνόκ. Σίγουρα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και πλούσια, θέτοντας μάλιστα και ζητήματα και ερωτήματα. Την προτεραιότητα έχει η αίθουσα. Ποιος έχει ερωτήσεις να υποβάλει. Σας υπενθυμίζω όμως ότι η Επιτροπή μας είναι πολύ ισορροπημένη όσον αφορά την ισότητα των φύλων, ε, να το ξέρετε. Ήμασταν τέσσερις άντρες και τρεις γυναίκες πριν φτάσει εδώ, κυρία Στυλθέ. Για να δείτε δηλαδή ότι είμαστε έτοιμοι για αυτά που λέτε. Λοιπόν, ποιο ε, θα δώσει τον ακτήριο λάκτισμα, ποιο έχει την πρώτη ερώτηση. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Παρακαλώ, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Σας άκουσα Διάβασα τα συμπεράσματα που υπάρχουν στην έκθεση. Έχω μία ερώτηση, λοιπόν. Πώς θα τα καταφέρουμε. Είμαι από την Ολλανδία και ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε τη συζήτηση για το κατά πόσο έχει χρησιμότητα η αναπτυξιακή βοήθεια. Τελικά. Από 0,8 πήγαμε στο 0,7 όσον αφορά το κομμάτι αναπτυξιακής βοήθειας στον προπολογισμό μας. Είμαστε και εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η συζήτηση οπότε υπάρχει κατά πόσο θέλουμε να τη δίνουμε αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια. Εσείς μιλάτε για την επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή. Είναι μια αρχή η οποία είναι μια αρχή που τη θέλετε και που και μας μας αρέσει. Εμείς δεν θέλουμε να αφισβητηθεί η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή, το ODA, αλλά τώρα ο ένας ή ο άλλος υπουργός από εδώ από εκεί κάθε τόσο στέλνει μια επιστολή στον ΣΑΣ, στην Αρμόδια Επιτροπή και λέει ας το συζητήσουμε. Εμείς λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα θα πείσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα όπως είναι η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή και για το κλίμα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Γιατί αν θέλουμε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση και λέτε εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, τότε πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Πώς θα πείσουμε τον κόσμο πρώτα απ' όλα να τηρήσει το ποσοστό για την επίσημη αναπτυξιακή αερογή και μετά να περάσει και σε ένα δεύτερο σύστημα αρρωγής για το κλίμα. Θέλετε να απαντήσετε τώρα αμέσω, ρωτά ο πρόεδρο. Ναι, αλλά δεν έχει μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ναι, φυσικά και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη βέβαια, Έχω την αίσθηση, κοιτάξτε δεν είμαι βέβαια εξοικειωμένη με το τι συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τις κάτω χώρες για παράδειγμα, η οποία είναι μια από τι λίγε χώρε, η οποία αν μη τι άλλο το έφτασε αυτό το 0,7% το στόχο και μπορεί να το μείωσε, αλλά κάποια στιγμή και έφτασε στο 0,7, αλλά η Γερμανία για παράδειγμα, η... ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας αυξάνει τον DCI. Οπότε υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν φτάσει στο 0,7%. Πάντως το ζήτημα όντως είναι ζωτική σημασία όπως το θέτετε. Και δεν έχω απάντηση, εννοείται. Αλλά για τη χρηματοδότηση ε, του κλίματος, το κλίμα βλέπετε είναι ο κύριος παράγοντας που μπορεί να κινητοποιήσει σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο γιατί η διεθνής κοινότητα παρατηρεί τι γίνεται. Η συζήτηση λαμβάνει χώρα. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα καθορίσουμε την προσθετικότητα, αν θα διασφαλίσουμε μια νέα χρηματοδότηση. Υπάρχει συμβουλευτική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ προκειμένου να βρεθούν τα 100 δις αμερικανικά δολάρια έχουν γίνει αναλύσεις. Βέβαια, το ζωτικό θέμα είναι πώς θα τεθεί σε εφαρμογή. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, γίνεται. Πολλά βέβαια από αυτά τα μέτρα είναι αλήθεια ότι χρειάζονται εφαρμογή σε διεθνές επίπεδο. Αλλά αν μιλάμε για τον φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, ακούμε ότι αυτό είναι εφικτό μόνο εφόσον συμφωνηθεί διεθνώς. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα, για παράδειγμα ο φόρος στο χρηματιστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, που σημαίνει ότι ακόμα και σε εθνικό επίπεδο μπορεί να υπάρχει μια προσέγγιση. Για παράδειγμα, στην Ευρωζώνη μόνο θα μπορούσε να γίνει κάτι. Δυνατότητες υπάρχουν. Ή στο σύστημα ε, αγοροπολισίας ε, εκπομπών. Δεν είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην ευρωπαϊκή βιομηχανία οι φόροι για το δεξίδιο του άνθρακα. Επίσης αποτελούν δυνατότητα για ανανέωση. Συνεπώς μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα τελικά κάτι τέτοιο. Είναι περισσότερο θέμα πολιτικής βούλησης και θάρρους, θάρρους αυτό κυρίω. Εγώ δουλεύω στον ίδιο τομέα που δουλεύετε κι εσείς. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε άλλου ανθρώπου. Ακούγονται διάφορες ανησυχίες για το πώς η αναπτυξιακή βοήθεια, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς τελικά ε, χρηματοδοτείται περισσότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Και εγώ έχω τις ίδιες ανησυχίες με εσάς, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, να πιέζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και να βάζουμε τα ίδια θέματα στο τραπέζι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο πώς θα πάτε αύριο στον Υπουργό Οικονομικών σας και θα τον πείσετε με τα σωστά επιχειρήματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ο χρόνος πιέζει. Ο κύριος Σέρενσον 11 και 40 ε, πρέπει να αποχωρήσει, οπότε έχουμε ήδη καθυστερήσει. Γι' αυτό θα έλεγα να ακούσουμε όλες μαζί τις ερωτήσεις. Ο κύριος Νόιζερ, η κυρία Ντεκέιζερ στη συνέχεια και μετά θα απαντήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε όλες τις ερωτήσεις. Στο μεταξύ δεν ξέρω μήπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, πριν την τελική απάντηση ή μετά. Μετά, ε, εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο εδώ. Λοιπόν, κύριε Νόιζερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ <clears throat> για την παρουσίαση της μελέτης η οποία διευκρίνησε ότι χρειαζόμαστε επιπρόσθετους πόρους για την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά παρουσιάσατε όλες τις ε, απόψεις και εγώ που προσπαθώ να εφαρμόσω στην πράξη αυτές τις ιδέες ε, η παρουσίασή σας ε, μου φάνηκε πολύ περίπλοκη γιατί βάλατε το στόχο του 0,7% που πολλές χώρες δεν έχουν επιτύχει και νομίζω ότι είμαστε ακόμη στο πρώτο βήμα. Τα επιπρόσθετα είναι α, επιπρόσθετη πόρη. Ε, παρουσιάστε μία εναλλακτική λύση ότι μπορεί κανείς να κάνει διπλοεγγραφές σε διάφορες περιπτώσεις. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι ευχαρίστως θα κάνουν τα κράτη-μέλη γιατί τους δίνουν διαπραγματευτική ικανότητα και μπορεί να τους απομακρύνει από την πραγματική επιτυχία των στόχων. Οπότε είπατε ότι έχουμε το στόχο του 0,7% και την υποχρέωση να συμβάλλουμε στην προστασία του κλίματος και όλα τα άλλα είναι ε, στόχοι που πρέπει να επιτύχουν την προστασία του κλίματος. Θα μου πείτε όμως τώρα πόσο θα μπορέσουν όλα αυτά να κατανεμηθούν και να φτάσουν στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Ευχαριστούμε κύριε Δεκαϊζέ. Άκουσα κι εγώ πολύ προσεκτικά την παρουσίασή σας που ήταν πολύ συγκεκριμένη. Αλλά κι εγώ όπως και ο Νόρμπερτ θα έλεγα ότι Μιλάτε κυρίως για πολιτικό θάρρος και πολιτική βούληση. Μα η οικονομική διακυβέρνηση έχει φέρει τεράστιους περιορισμούς στις χώρες μέλη. Τους έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Οπότε είναι περισσότερο θέμα πολιτικής βούλησης ε, παρά ε, στραγγαλισμού Πέρα λοιπόν από αυτό το 0,7% τι σημαίνει. Σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά όποια επιλογή και αν διαλέξετε σελίδα 13 περισσότερα που θα τα βάλετε στον λογαριασμό στον άλλο με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ένα είναι το ζητούμενο, περισσότερα χρήματα. Οπότε, πού θα τα βρείτε. Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, αναφερθήκατε και την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να είναι μια λύση σύμφωνη, αλλά το ερώτημα είναι αυτό, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Γιατί το κατά πόσο οι πολιτικοί θα το δεχτούν ή θα το δεχτούν εξαρτάται από το πού θα βρεθούν τα χρήματα, ποιε θα είναι οι πηγέ χρηματοδότηση. Γιατί έτσι κι θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα. Άρα κάπου πρέπει να βρεθούν. Οπότε η συζήτηση πρέπει να γίνει για τι πηγέ χρηματοδότηση. Πολύ περισσότερο παρά να μιλάμε για το θάρρο που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί και οι χώρε. Πρόεδρο, πολύ σωστά. Ναι. Απαντήστε μα παρακαλώ. Μετά είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πάρει το λόγο, έτσι. Εκτός μικροφώνου πάλι ομιλήτρια. Δεν την ακούμε. Μικρόφωνο. Ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια. Το σωτική σημασία ε, ερώτημα, το από πού θα έρθουν τα χρήματα, δεν ήταν στο κέντρο όντω τη παρουσίασή μου. Θα το θίξω όμω. Και θέλω να αναφερθώ στους, ε, στην έκθεση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναφέρεται και κάπου και στο κείμενο. Στην παρουσίαση πρέπει να το είδατε ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ανάλυση για το από πού θα μπορούσαν να προέλθουν τα κονδύλια. Και κατέληξε στο ότι μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι εφικτό. Οι περισσότεροι πόροι θα ερχόντουσαν από το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με αυτό το σύστημα αδειών εμπορίας δηλαδή, από τον φόρο χρηματοστοπικών συναλλαγών και ίσως και από την εισαγωγή κάποιου φόρου για το διοξίδιο του άνθρακα. Δυνατότητες λοιπόν υπάρχουν και αναφέρονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις γνωρίζει και η Επιτροπή τις έχει καταγράψει. Συνεπώς είναι περισσότερο θέμα εφαρμογής τους και όχι κατά πόσο υπάρχουν ή όχι. Υπάρχουν. Αλλά όντω είναι ε, θέμα ζωτική σημασία. Τώρα για το στόχο του 0,7%. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι αυτό που μπορεί περισσότερο να κινητοποιήσει η χρηματοδότηση είναι ακριβώς το κλίμα. Σε πολλές χώρες δεν έχει επιτευχθεί το 0,7%. Όμως, τώρα που υπάρχει ο παράγοντας κλίμα, πιστεύω ότι η συζήτηση παίρνει άλλε διαστάσει. Γίνεται πιο ζωντανή από ό,τι όταν συζητούσαμε για την επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή. Α μην πούμε να πετύχουμε πρώτα το 0,7% παντού και μετά θα δούμε. Όχι. Η χρηματοδότηση για το κλίμα επήγει τόσο πολύ, ακόμα και για αναπτυξιακά θέματα, που δεν μπορεί να περιμένει. Το θέμα του κλίματος θα επηρεάσει αρνητικά πάρα πολλά επιτεύγματά μας. Συνεπώς, η χρηματοδότηση αυτή για το κλίμα είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε παράλληλα με την ανάπτυξη. Η συζήτηση αυτή δεν πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό και μιλάμε για την ολοκλήρωση. Πιστεύουμε ότι τα δύο, η ανάπτυξη και το κλίμα, πάνε μαζί, αποτελούν ένα. Όντως είμαστε σε μια κρίση η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και γι' αυτό και προσπάθησα στον ορισμό μου εντό αγωγικών να πω ότι θα μπορούσε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα να υπήρχε διπλή εγγραφή. Είναι ένα συμβιβασμό. Ακριβώ επειδή υπάρχει οικονομική κρίση. Αν δεν υπήρχε, θα έλεγα 0,7 συν. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει η οικονομική κρίση, γι' αυτό και θα επέτρεπα αυτή τη διπλή εγγραφή για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Αυτά. Πρόεδρος, ναι, απαντήσατε πλήρως. Το λόγο τώρα τον έχει ο κύριος Στέφαν Ναγκδινέ. Ελπίζω να μην ε, έσφαξα πολύ το όνομά σας, όπως το πρόφερα, αλλά μπορείτε να το επαναλάβετε εσείς σωστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στεφάνα Νιέ. Στα αγγλικά θα μιλήσω, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο και που μας προσκαλέσατε εδώ στην παρουσίαση αυτή. Πρώτα απ' όλα, θα χρειαστούμε περισσότερη χρηματοδότηση για το κλίμα για να πετύχουμε την, ε, τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών. Η χρηματοδότηση πρέπει να έρθει από διάφορες πηγές, δημόσιο, ιδιωτικό, τομέα, ε, καινοτομία. Υπάρχει η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή και υπάρχει για το θέμα της προσθετικότητας. Η προσθετικότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η χρηματοδότηση που δίνεται, δίνεται παραπάνω από ένα ποσό. Και ποιο είναι αυτό το ποσό όμως. Και εδώ ακριβώς είναι που δεν συμφωνούν οι διάφορες πλευρές και είναι δύσκολο να επιτευχθεί συνένεση. Παρ' όλα αυτά, στην έκθεση Monterey κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στη χρηματοδότηση του κλίματος και τη χρηματοδότηση για άλλους αναπτυξιακούς σκοπούς. Αν κοιτάξετε την έκθεση που είναι του 2011, θα δείτε ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει πάνω από ένα όριο, που είναι ο μέσος όρος του ODA, της επίσημης αναπτυξιακής αρρωγής δηλαδή, έτσι όπως αυτή είχε το 2009. Τι ακριβώς είναι η επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή. Υπάρχει ορισμός. Είναι η χρηματοδότηση που δίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και η χρηματοδότηση αυτή δίνεται για διάφορους σκοπούς. Μπορεί να δοθεί για δράσεις στον τομέα του κλίματος, αλλά και για άλλες δράσεις. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε εδώ για διπλή εγγραφή όταν χρησιμοποιούμε χρήματα από την επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή για το κλίμα. Γιατί είπαμε υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και αυτές ισχύουν και για την περίπτωση του κλίματος. Το σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει διαφάνεια για το πού πηγαίνουν τα χρήματα τη επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή, κατά πόσο χρηματοδοτούν άλλε προτεραιότητε, την ανακούφιση από τη φτώχεια, για παράδειγμα, ή την εκπαίδευση, την υγεία. Βέβαια, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και πολλές γκρίζε ζώνες και φαίνεται αυτό και στην έκθεση, γιατί υπάρχουν όντως κοινά ωφέλη ε, από τη χρηματοδότηση του κλίματος στην ανάπτυξη και από την ανάπτυξη στο κλίμα. Φυσικά, τα δύο ε, εντάσσονται πλήρως στην αναπτυξιακή μας πολιτική απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και γι' αυτό και γίνεται ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση τώρα που έχουμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, στις προτάσεις δηλαδή που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές. Γιατί πράγματι υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο μιλάμε για την χρηματοδότηση του κλίματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται επενδύσεις προκειμένου να αντισταθούμε στις αλλαγές του κλίματος. Από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχουν και καθαρές τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Για να ολοκληρώσω. Στην πράξη έχουμε εφαρμόσει μια συγκεκριμένη αρχή για να ορίσουμε τη χρηματοδότηση του κλίματος σε σχέση με την γενικότερη αναπτυξιακή χρηματοδότηση έτσι όπως αυτή περιλαμβάνεται στην έκθεση του Μοντερέι. Φάνηκε όμως ότι υπάρχουν δυσκολίες και από αυτή τη συζήτηση, γιατί αντί να επικεντρωνόμαστε στις λεπτομέρειες για τις διάφορες ε, έννοιες της προσθετικότητας, καλύτερα θα ήταν να κοιτάξουμε πού θα βρούμε τους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε την ε, αντίσταση στις κλιματικές αλλαγές. Τα σχόλια από τους ευρωβουλευτές εδώ έδειξαν ότι αυτό ακριβώς είναι και αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εμείς βασιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στηρίξει την κινητοποίηση περισσότερων πόρων για τη χρηματοδότηση του κλίματος και από τους δημόσιους προϋπολογισμούς αλλά και από άλλους πόρους. Τελικά και από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί όχι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αυτό το τελευταίο είναι για μένα και το συμπέρασμα και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Εσεί τι ζητήσατε, ζητήσατε να μπορείτε να βασιστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα πάντα μπορείτε να βασίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε οι πρώτοι που καταδικάζουμε ε, τη διπλή γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις σημερινές ανάγκες. Προσπαθούμε να υπάρχει συνοχή στη συζήτησή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δικιά της την πλευρά, ε, και αυτή είναι μεταξύ σκυλες και χάριδος, κακά τα ψέματα δεν ε, απέφυγε να κάνει τη διέκριση ανάμεσα στα χρήματα που πηγαίνουν για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές από τη μια και την ανάπτυξη από την άλλη. Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν γνωρίζουμε τελικά ποια είναι τα ποσά τα οποία άλλαξαν ε, προορισμό. Γιατί υπάρχει αυτό και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να το γνωρίζω αυτό, να ξέρω δηλαδή τι ποσά αρχικά ήταν για να πάνε στην επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή και τελικά πήγαν σε άλλους προορισμούς, ε, συναφείς βέβαια βάση του ΩΣΑ, αλλά πάση περιπτώσει όχι ακριβώς αυτούς, συναφείς. Αυτό που μας κάνει να βγαίνουμε έξω από τα ρούχα μας εδώ είναι ότι πολλές χώρες αδιαφορούν πλήρως αφήνουν να γίνεται η συζήτηση και διαφορούν πλήρω. Η Επιτροπή πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να βασιστεί σε μας. Μπορεί να φωνάζουμε, αλλά είμαστε ενωμένοι και φωνάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση, αν μη τι άλλο. Κατόπιν αυτών, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για αυτό το θέμα και συνεχίζω για να σας εισαγάγω στο επόμενο θέμα. Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας σήμερα το πρωί είναι ο κύριος Κλάου Σόρενσον. Τον υποδεχόμαστε εδώ, είναι τιμή για μας. Πρόκειται για τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ. Πριν από ένα μήνα, κύριε Σόρενσεν, ήσασταν εδώ μαζί μας πάλι για να μας ενημερώσετε όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία. Δυστυχώς, τον τελευταίο μήνα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Σήμερα βρισκόμαστε σε σύραξη και μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε δει ε, πολλές, ε, πολλά ρεπορτάζ για θύματα, πολλοί άριθμα θύματα, τα οποία έχουν σφαγιαστεί ψυχρό. Τώρα λοιπόν θέλουμε να ακούσουμε από εσά. Τι δράσεις έχουν αναλάβει οι δωρητές με ανθρωπιστική βοήθεια και επιπλέον θέλουμε να μας ενημερώσετε και για άλλες περιπτώσεις ανθρωπιστικής αρρωγής στις οποίες εμπλέκεται η ΕΚΟ για να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Τζόρτζ Όκοτ Όμπο που είναι ο διευθυντής του Αφρικανικού Γραφείου της Υπατης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι από την Ουγγάντα, είναι δικηγόρος με μεγάλη καριέρα στα Ηνωμένα Άθνη. Προηγουμένως, πριν αναλάβετε τα τελευταία σα καθήκοντα, ήσασταν ε, διευθυντής για την διεθνή προστασία. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε από εσά να μας εξηγείτε τι ακριβώς κάνει η Πατερμοστή των Ηνωμένων Εθνών για να ανακουφίσει στην περίπτωση διαφόρων κρίσεων στην Αφρικανική Ήπειρο, μεταξύ των οποίων εκείνη στο Σαχέλ, στο κέρα τη Αφρική, αλλά επίση και στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν. Εσείς κύριε Σόρενσον, θα ήθελα να ξεκινήσετε παρουσιάζοντάς μας το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τις συνεχείς ανθρωπιστικές κρίσεις στην Αφρική αλλά και όχι μόνο. Να μας μιλήσετε και για τη Συρία και την Ιεμένη. Και μετά ο κύριος Σοκοτ Όβου μπορεί να πάρει τη σκητάλη από εσά και να συμπληρώσει με άλλες πληροφορίες όσον αφορά την οπτική γωνία των Ηνωμένων Εθνών. Μετά φυσικά θα υπάρξει περιθώριο για ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Σέρενσον. Για 10-15 λεπτά είναι εντάξει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό είναι να ξεκινήσουμε με τη Συρία, γιατί σε καθημερινή βάση τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ο κ. Λατσούς που είναι υπεύθυνος των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνευτικές ε, ε, αποστολές ε, έχει δώσει την περιγραφή για την κατάσταση που επικρατεί εκεί σαν κάτι το οποίο πλέον είναι πολύ κοντά στον πλήρη εμφύλιο πόλεμο. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Και όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό, ήδη από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, είχαμε δει τεράστιους αριθμούς εσωτερικά εκτοπισμένων πολιτών, γυναικών, παιδιών που είχαν πυροβοληθεί Υπάρχει έλλειψη παροχής νερού, υπάρχουν προβλήματα με τα φάρμακα, έχουν κλείσει τα σχολεία. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν πια στα σχολεία, τουλάχιστον όπως το έκαναν πριν. Και πάνω λοιπόν από τα άμεσα προβλήματα που έχουμε, η κατάσταση αυτή δεν υπόσχεται τίποτα καλό για το μέλλον, γιατί αν τα παιδιά δεν πάνε σχολείο ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρουμε ε, πού θα στραφούν για να εμπνευστούν τις ιδέες τους, την ιδεολογία τους κτλ. Ήμασταν ιδιαίτερα δραστήριοι βέβαια στο επίπεδο το καθαρά ανθρωπιστικό. Δεν χρειάζεται να πει κανείς βέβαια ότι το ανθρωπιστικό στοιχείο δεν θα λύσει το πρόβλημα. Απαιτεί πολιτική δράση, απαιτεί ίσως κάτι περισσότερο από πολιτική δράση, δεν είναι δική μου δουλειά αυτό, αλλά εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον σε επίπεδο ανθρωπιστικό να βοηθήσουμε και εμπλεκόμεθα με όλους όσους συμμετέχουν. Προέρχομαι από, ένα, μια πρωινή συνάντηση με τον κύριο Κίλι Μπέργκερ, ο οποίος είναι υπεύθυνος των Ηνωμένων Εθνών εκεί σε επίπεδο ανθρωπιστικό και τον, του Ερυθρού Σταυρούση μάλλον ε, κρατιούνται στη Συρία, έχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνεργατών πάντα μέσα στη Συρία και να είμαι ειλικρινής υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού, για τη δυνατότητα πρόσβασης, για το αν μπορεί ε, η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ να είναι εκεί δραστήρια. Απαιτούνται δράσεις και αναλαμβάνονται δράσεις, δράσεις οι οποίες ε, πολλές φορές ε, διεξάγονται υποχρεωτικά χωρίς κάποια αδειοδότηση επίσημη και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, ακόμη και προβλήματα πολιτικού τύπου. Σε επίπεδο ανθρωπιστικό λοιπόν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Ο υπεύθυνο των Ηνωμένων Εθνών είναι υπεύθυνο για την περιοχή, αλλά έρχεται κυρίως σε επαφή με την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση παραμένει και ο Orchard λοιπόν έρχεται σε επαφή μαζί τους, διότι ελέγχουν χωρικά την περιοχή. Ενθυμίστε ίσως ότι όταν είχαμε το τελευταίο φόρουμ το ανθρωπιστικό για τη Συρία εδώ και τρεις εβδομάδες στη Γενέβη, συνέβη αυτό το οποίο συνέβη ε, και τώρα. Την τελευταία στιγμή οι Σύριοι ε, κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Υποτίθεται ότι συνυπογράφουν το πρόγραμμα ανταπόκρισης το οποίο τους προτείνονται και το οποίο είχαν αρνηθεί μέχρι τότε να υπογράψουν. Την τελευταία στιγμή το υπέγραψαν. Βέβαια εμείς τους πιστέψαμε αλλά και δεν τους πιστέψαμε. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί ε, το πρόγραμμα αυτό, να διευκολυνθούν οι θεωρήσεις, να ανοίξουμε γραφεία τα οποία δεν είχαν αδειοδοτηθεί, πότε θα αδειοδοτηθούν τα γραφεία, να μην παρεμποδίζουν τα τρόφιμα και τα υλικά και τους εξοπλισμούς που μεταφέρουμε στην χώρα αυτή. Περιμένουμε νέα λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Εγώ ο ίδιος Έχω δημιουργήσει ένα σύνδεσμο ανάμεσα σε αυτές τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρξουν και στην δυνατότητά μας να αυξήσουμε την ένταση των προσπαθειών μας. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα αν ταυτόχρονα δημιουργούνται ε, τροχοπέδες και εμπόδια στην προσπάθεια επίδοσης, θα έλεγα, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα νέα από τη χώρα είναι, θα έλεγα, δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα. Η κυβέρνηση σε ορισμένους τομείς της θεωρήση, σαν παράδειγμα, εκδίδει κάποιες βίζες, δείχνει κάποια καλή βούληση, από την άλλη πάλι βέβαια δυστυχώς δεν παίρνει τα μέτρα τα οποία απαιτούνται το αντίθετο και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι πού θα φτάσουμε. Δεν μπορούμε εμείς να παρετηθούμε, δεν μπορούμε εμείς να φύγουμε από τη Συρία, πολύ απλά. Γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι και οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τη βοήθειά μας. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να βρούμε μάλλον έναν διαφορετικό τρόπο για να πιέσουμε την κυβέρνηση της Συρίας, να τους θέσουμε ενώπιον των ευθυνών τους έτσι ώστε να μας πούν με ποιο τρόπο έχουν ανταποκριθεί μέχρι τώρα σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπογράψει. Και όταν είχε έρθει εδώ η Βάλερη Έιμος, συζητήσαμε ε, το θέμα της επανασύγκλησης του Φόρουμ του Ανθρωπιστικού για τη Συρία έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ε, ένα ελάχιστο επίπεδο πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση. Βέβαια, το θέμα δεν είναι μόνο ποσοτικό. Εμείς από πλευράς μας της ΕΚΟ χρησιμοποιούσαμε το λειτουργικό μας απόθεμα, χρησιμοποίησαμε 10 εκατομμύρια και μετά άλλα 10 εκατομμύρια Τώρα είμαι σε συνομιλίες με τις υπεύθυνε ε, υπηρεσίες της Επιτροπής, τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε κάποια επιπλέον χρήματα ε, για το απόθεμα ε, εκτάκτων καταστάσεων. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι έτσι ώστε να μην μείνουμε από λεφτά και θέλω και κάποιες διαβεβαιώσεις έτσι ώστε αυτά τα οποία υποσχόμεθα να μπορούμε να τα παραδώσουμε γιατί αλλιώς τι νόημα έχει. Υπάρχει ανάγκη χρημάτων λοιπόν, υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι άνθρωποι που θα πρέπει να υποστηριχθούν και το θέμα είναι βέβαια να μας δοθεί και πρόσβαση για να χορηγήσουμε τη βοήθεια αυτή. Είμαι σε επαφή και με την Ερυθράη Μισέλινο της Συρίας, τον δόκτορα Ατάρ αν γνωρίζετε. Ο δόκτορ Ατάρ κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, προσπαθεί να εξισορροπήσει από τη μία τα της κυβέρνησης και από την άλλη τις ανάγκες του λαού του. Πάρα πολλοί έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πλέον Κάποιοι από αυτούς ε, δυστυχώς θυσιάστηκαν ήδη και ο Κίλεμπεργκερ μου είπε σήμερα ότι η Ερυθράη ημισέλινος θα ήθελαν το ΣΑΚ, η υπηρεσία αυτή χορήγησης βοήθειας, να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές τους και πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει επιπλέον ε, την προσπάθεια αυτή. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε τώρα στα 20 εκατομμύρια. Αν προσθέσουμε και αυτά τα οποία έχουν ήδη υποσχεθεί τα κράτη-μέλη, φτάνουμε τα 32 εκατομμύρια και υπάρχουν και κάποια επιπλέον χρήματα από τον ε, προϋπολογισμό ανάπτυξης, 23 εκατομμύρια και θα επανέλθω σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε περισσότερες πιστώσεις. Απαιτείται να πιέσουμε όμως και μας στηρίζει το σύνολο της ε, κοινότητας της διεθνούς. Η εμένη μας ανησυχεί επίσης. Είναι λίγο εκτός ραντάρ γιατί ήταν τα πράγματα πολύ άσχημα, μετά ξέσπασαν άλλες κρίσεις όπως η Συρία, το Μαλί κτλ και την ξεχάσαμε λιγάκι. Έφυγε λίγο από την οθόνη μας. Πάντως να σας πω ότι ένα εκατομμύριο παιδιών υποφέρουν από έντονη ασυτεία. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό μπορεί να είναι αυτό γιατί μπορεί να πάθουν εγκεφαλικές βλάβες, κάτι το οποίο δεν είναι ανακτήσιμο και θα έχουμε μια ολόκληρη γενιά γιατί θυμίζω ότι 10 εκατομμύρια οι εμενίτες ζουν κάτω από πλήρη τροφιμική ανασφάλεια και προς τα εκεί έχουμε δώσει χρήματα. Έχουμε κάποιες δυνατότητες πρόσβασης στην περιοχή της Ιεμένης. Κατά κάποιο τρόπο εποφελούμεθα από την καλή, από τις καλές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί μετά από την επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτιέρες και του δικού σας ε, αφεντικού σε εισαγωγικά και της δικής μου, της ε, κυρίας Γεωργίεβα. Έχει δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα και μας επιτρέπουν να χορηγούμε την βοήθειά μας στην επισητιστική. Αλλά έχουμε και εδώ ανάγκη από κάποια επιπλέον χρήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβεώσουμε στην περιοχή αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου. Το θέμα είναι η επισητιστική βοήθεια να παραμένει γραμμικά διαθέσιμη και να μην στερέψει στη μέση της διαδικασίας. Για το Σουδάν τώρα και το Νότιο Σουδάν. Λυπάμαι γιατί έρχομαι εδώ και σας δίνω όλα τα κακά νέα. Ε, δεν είναι το στυλ μου αυτό. Εγώ είμαι αισιόδοξο άνθρωπος, αλλά όταν τα βλέπει όλα μαζί τα πράγματα πάνε άσχημα. Λοιπόν, ελπίζαμε στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν ότι θα συμφωνούσαν στο τέλος του 11 ε, για τα εισοδήματα του πετρελαίου που προέρχονται από πετρέλαιο. Δεν ξέρω ποιος πυροβόλησε τον άλλο ή ποιος αυτοπυροβολήθηκε. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό και το πρόβλημα είναι ότι το 90% του προϋπολογισμού του Νοτίου Σουδάν προέρχεται από το πετρέλαιο, την εξόριξη πετρελαίου. Ε, ε, γι' αυτό λοιπόν θέλουν τώρα να καταστήσουν τους αντάρτες που είχαν δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι βέβαια όταν δεν πληρώνονται με το μισθό τους κάνουν άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουμε μπροστά μας μια νέα προοπτική ενός αποτυχημένου κράτους, ενός κατεστραμμένου κράτους ή ήδη έχει ε, υπάρξει ένα κατεστραμμένο κράτος, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω καταστροφικά προβλήματα. Στο Βόρειο Σουδάν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συστηματικά δεν σέβεται τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές, προσπαθούν να εθνικοποιήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια, Ακόμα και οι φίλοι μας από τον Ευηθρό Σταυρό έχουν τεράστιες δυσκολίες για να έχουν πρόσβαση στις βάσεις τους. Υπάρχει επίσης και το κύμα των προσφύγων, υπάρχουν και οι απάτριδες οι οποίοι ουσιαστικά πιέζονται προς τον Άνω Ήλο, μετά καταλήγουν στο Νότιο Σουδάν και στο τέλος σε στρατόπεδα προσφύγων της Τζούμπα. Η κατάσταση λοιπόν χειροτερεύει. Οι αριθμοί επίσης μεγαλώνουν και σε αυτή τη φάση αρχίζει η εποχή των βροχών. Είμαστε στην εποχή των βροχών, οπότε είναι και δύσκολο να πάνε ε, τα τρόφιμα. Βέβαια το καλό είναι ότι εμείς είχαμε ήδη τοποθετήσει αρκετά τρόφιμα μέσω του Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφής, Τροφίμων, Είχαμε τοποθετήσει ε, τρόφιμα στην χώρα σε συγκεκριμένα μέρη, επί τη βάση όμως των αναγκών που είχαν προβλεφθεί πριν 4-5 μήνες, κάτι το οποίο δεν αρκεί σήμερα. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα λοιπόν. Και εδώ θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αυξηθεί η βοήθεια που δίδουμε για τις χώρες αυτές για το Σαχέλ, κυρία Στίφλερ, ήσασταν εκεί χθε. Είδατε ότι το θέμα του λοιμού αντιμετωπίζεται με ικανό θα έλεγα τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλους δωρητές. Δεν θέλω να αυτοσυγχαρώ να, τις υπηρεσίες μου αλλά παρόλα αυτά στην περίπτωση του ΣΑΕΛ λειτουργήσαμε κάπως πιο προληπτικά. Περισσότερο από ό,τι κάναμε στο κέρας της Αφρικής. Στο κέρας της Αφρικής δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε σωστά, αλλά αυτή τη φορά προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την παρουσία μας. Έχουμε σωστό διάλογο με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, προκαταβάλουν τις πιστώσεις που έχουν στη διάθεσή τους και υπάρχει αυτό το desk για το Σαχέλ το οποίο στην ουσία προσπαθεί να ενισχύσει τις τοπικές κοινότητες έτσι ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη αυτού του φαινομένου. Όλα αυτά λοιπόν μου δίνουν κάποιες ελπίδες. Αυτό που δεν μου δίδει ελπίδες είναι η χειροτέρευση της πολιτικής κατάστασης. Γιατί όσο προσπαθούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί συνδυάζοντας την αναπτυξιακή βοήθεια με την ανθρωπιστική βοήθεια, έτσι ώστε να σταθούν στα πόδια τους οι κοινότητες και να βγουν σιγά σιγά από την κρίση με λίγη βοήθεια στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής βοήθειας, των σχολείων. Δυστυχώς όμως η πολιτική κατάσταση στην περιοχή χειροτερεύει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ με λεπτομέρειες στο Μαλί, όπου ο βορράς του Μαλί είναι αποκλεισμένος για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το μόνο φως, μικρό φως ελπίδας που έχουμε είναι ότι η Βάλερη Έιμος έχει διορίσει ένα πολύ ικανό ε, συντονιστή στα ανθρωπιστικά για το Σακέλ και τώρα έχει αρχίσει να προσπαθεί να βρει τρόπους έτσι ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των κομμάτων και των εμπλεκομένων στην περιοχή έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα πρόσβασης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Έχουμε ικανότητε και έχουμε κάποια περιθώρια οικονομικά σε αυτή τη φάση. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές αυτές σε ένα περιβάλλον περίπλοκο και επικίνδυνο. Η αστάθεια δεν αφορά μόνο το Σαχέλ, αλλά και την Βόρεια Νιγηρία και τη Βυτική Νιγηρία. Εκεί έχουν υπάρξει αρκετά προβλήματα, αλλά δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Για το κέρας, για μια ακόμη φορά, ξέρετε την πρωτοβουλία Share που έχουμε ξεκινήσει, όπως ακριβώς και με την πρωτοβουλία Azir ΣΑΧΕΛ, δράση στο Σαχέλ προσπάθεια συνδυασμού της ανθρωπιστικής βοήθειας με μια εξαιρετική στρατηγική που θα επιτρέψει στις περιοχές όπου υπάρχει σχετική ειρήνη και πρόσβαση να δημιουργήσουμε κάποια στοιχεία ελπίδας. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους διεθνείς δωρητές, ιδιαίτερα τους Αμερικανούς που είναι δραστήριοι στην περιοχή αυτή εμείς είπαμε ότι βάλτε τους δικούς σας διοικητικούς υπαλλήλους να ασχοληθούν με την περιοχή αυτή. Εμείς θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας περισσότερο στο Σαχέλ, αλλά οι μεν θα στηρίζουμε τους δε. Και ελπίζουμε ότι στο τέλος θα υπάρξει μια ουσιαστικά κοινή βοήθεια για την αύξηση της αντοχής των κοινοτήτων, κάτι το οποίο επιδιώκουμε και για το Σαχέλ και για το κέρας της Αφρικής. Μπορώ να συνεχίσω χωρίς να σταματήσω ποτέ, δεν θα ήταν δίκαιο. Can go on and on. Ξέρουμε ότι μπορείτε να ε, συνεχίσετε, αλλά θα δώσω μέσω στον λόγο στον κύριο Κώτη για 10 λεπτά, διότι στη συνέχεια υπάρχουν τόσες ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές οι οποίοι μας υποδέχτηκαν. Ο κύριος Σόρενσεν έχει διευκολύνει πολύ το έργο μου γιατί τα τρία θέματα τα οποία ήθελα να σχολιάσω για το κέρας της Αφρικής και το Μαλί μας παρουσίασε ποιο είναι το δράμα που αντιμετωπίζουμε οπότε θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω περισσότερο χρόνο για να απαντώ σε ερωτήσεις σας. Όσον αφορά το κέρας της Αφρικής πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή αυτή όπου υπάρχουν νέα κράτη και 108 εκατομμύρια κατοίκους είναι η σκηνή ε, μεγαλύτερων ε, πληγών και ε, δυστυχιών του, των λαών. Και αν πάρω ένα παράδειγμα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Σομαλίας, στην περιοχή αυτή και μόνο πέρυσι είχαμε 200.000 Σομαλούς που εκτοπίστηκαν σε 12 μήνες στην περιοχή αυτή και στους πρώτους μήνες αυτού του έτους είχαμε ακόμη 20.000 στη, εντός της χώρας ε, βλέπουμε ότι υπάρχει εσωτερική μετακίνηση 1,5 εκατομμυρίου από τα 7 εκατομμύρια. Υπάρχουν πολλοί ε, τοξικοί παράγοντες, είτε μιλάτε για την ξηρασία, για της ε, διενέξεις εάν μιλάτε για την τρομοκρατία και τα θέματα της ε, εσωτερικής ή διεθνούς ασφαλείας και έχουμε τους μεγαλύτερους, ε, τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις προσφύγων στην περιοχή. Βλέπουμε ότι έχουμε 500.000 σόλμαλους, 10.000 πρόσφυγες εκ των οποίων οι γονείς γεννήθηκαν μέσα στον καταβλισμό τον ε, προσφυγικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ε, ας μιλήσουμε τώρα για το Σουδάν και ιδιαίτερο στο Νότιο Σουδάν. Διότι αν σκεφτούμε κύριε Πρόεδρο ότι σήμερα στην αίθουσα αυτή είμαστε περίπου 50 άτομα και αν σκεφτούμε ότι τα 57 άτομα είναι 50 παιδιά που έχουν μετατοπιστεί από τον μπλε Νίλο ο και άλλες περιοχές προς το νότιο Σουδάν τότε ε, μέχρι να, φτάσουμε, να φτάσουν στον προορισμό τους θα είχαν πεθάνει τα μισά και αυτό συνέβη στο Σουδάν διότι όπως μας είπε ο κύριος Σόρενσεν αυτό που διαπιστώσαμε ε, στην απογραφή μεταξύ των δύο Σουδάν είναι ότι στις δύο αυτές περιοχές υπήρξαν μετατοπίσεις προς την Αιθιοπία και έχουμε εξ αυτών 140 στο Νότιο Σουδάν. Στις τελευταίες 10 μέρες και μόνο περίπου 50.000 άτομα μόνο σε 10 μέρες εκ των οποίων οι μισοί μετακινήθηκαν προς μία περιοχή και άλλοι προς κάποια άλλη. Και ε, υπάρχει επίσης ε, το πρόβλημα των επιδημιών, ευλογιάς, ε, χολέρας, και τέλος το τελικό θέμα είναι ακριβώς αυτό το οποίο έθιξε και ο κύριος Σόρενσεν, δηλαδή η κατάσταση στο Μαλί. Και εκεί οι αριθμοί δυστυχώς είναι πολύ ανησυχητικοί γιατί στην περίοδο από την αρχή του έτους περίπου 200.000 κάτοικοι του Μαλή έχουν μετακινηθεί προς την Μαυριτανία, τη, τον Ήγυρα και άλλες χώρες ε, και μετά άρχισε να βρέχει. Οι πρόσφυγες έχουν μόνο τέντες, αντίσκηνα, τα οποία παρέσυραν οι βροχές στον Ήγυρα και μπορούμε μόνο να ε, προσφέρουμε βασική και ε, ε, ελάχιστη βοήθεια και γι' αυτό είμαι εδώ. Ορισμένα από τα μηνύματα τα οποία θα σας απευθύνω όταν τελειώσω αυτή την παρουσίαση θα το εκφράσουν διότι είναι ζωές που κινδυνεύουν κύριε Πρόεδρε και είναι βασική αποκατάσταση των ζημιών και εντοχή αλλά εντός 30 λεπτών σε πολλές καταστάσεις στις πιο επίγουσες στο νότιο Σουδάν άνθρωποι πεθαίνουν μέσα σε μισή ώρα. Αυτό είναι σοβαρό και αυτό προσπαθεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε ο κύριος Όρενσεν και η ομάδα του να διατηρήσουμε εν ζωή τους ανθρώπους αυτούς και το δεύτερο είναι ότι μέσω εσάς θέλω να ευχαριστήσω τις χώρες σας διότι κάθε μία από αυτές με τον τρόπο της προσπάθησε να μας στηρίξει να δώσουμε ελπίδα και ευκαιρίες είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε διμερός και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Επίσης νέες ευκαιρίες πρέπει να δοθούν σε αυτούς τους περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που ε, εξέφρασα, των οποίων εξέφρασα την κατάσταση. Πολλοί είναι νέοι και ιδίω ε, άνδρες οι οποίοι ε, είναι στην περιοχή γύρω στο Αρσαντάμ, το ΑΚΕΜ είναι οργανώσεις οι οποίες απειλούν όχι μόνο την επιβίωσή τους αλλά ακόμη περισσότερα. Ορισμένοι από αυτούς σήμερα είναι στο Μαγκρέμπ εχμάλωτοι. Εάν δεν δώσουμε ευκαιρίες αυτούς τους νέους οι οποίοι είναι εις ε, την ε, ε, μπορούν να, στο οποίο μπορεί να επιτεθεί, να επιτεθεί ο στρατός. Θα δυναμητήσουμε λοιπόν όλες τις προσπάθειές μας εάν δεν αντιδράσουμε είτε διμερείς είτε πολυμερείς οι λύσεις οι πολιτικές οι πολιτικής οικονομίας θα προέλθουν από την επίλυση των θεμάτων σε αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ μετά από αυτές τις δύο ομιλίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ε, ουσιαστικές και συγκινητικές και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Σόρενσεν και τον Μπουρμέ και μιλώ για τον κύριο Σόρενσεν διότι γνωρίζουμε την ποιότητα της εργασίας του προγράμματος ΙΧΟ και έχετε μία γενική διεύθυνση για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Αλλά στο σύνολο των προβλημάτων και για να ακολουθήσω το σκεπτικό μου βεβαίως και θα εισακούσουμε τις σας. Αλλά σε όλα αυτά τα οποία μας είπατε, η δυσκολία και η παρέμβαση η οποία υπάρχει μεταξύ πολιτικών θεμάτων, θεμάτων αναπτύξεως, αμήνης και ανθρωπιστικών, όλα τα θέματα αυτά πρέπει να συμβαδίζουν και τελικά η λύση πρέπει να είναι πολιτική, περιμένοντας όμως την πολιτική λύση δεν πρέπει να πεθαίνουν οι άνθρωποι και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν δύο σημαντικότατες πτυχές σε αυτά που είπατε και είναι το εξής. Καταρχήν, η ανθρωπιστική πρόσβαση γιατί είναι το βασικό πρόβλημα. Αναφερθήκατε σε περιοχές του Μαλή, της Σομαλίας, στο Μπλε Νείλο, το Νότιο Κορδοβάν. Είναι περιοχές όπου υπάρχει δυσκολία να προσχωρήσει, να έχει πρόσβαση η ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, δεν μιλάμε για τον νήλο και άλλες ε, και μετά την πρόσβαση θα μιλήσω για την αποτελεσματικότητα. Καταρχήν όμως για τη Συρία κύριε Σόρενσεν. Εσείς μας είπατε ότι έχουμε δαπανίσει ή δεσμεύσει τόσα εκατομμύρια. Ξέρουμε τους Σύριους. Τους ξέρω και εγώ καλά και ορισμένοι άλλοι τους γνωρίζουν, λένε ναι, και μετά αρχίζουν τα εμπόδια και τραβάει η κατάσταση. Εάν λοιπόν δεσμεύσετε ακόμη περισσότερη χρηματοδότηση τώρα τι απέδωσε μέχρι τώρα η χρηματοδότηση αυτή. Μήπως εκεί θα έχουμε ορισμένα χρήματα τα οποία δεν θα αποδίδουν γιατί απλώς οι Σύριοι δεν τα θέλουν. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο. Επίσης δεν θα αναφερθώ σε όλα τα σημεία αλλά στο θέμα του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν. Ξέρουμε ότι το θέμα είναι πολιτικό. Βέβαια υπήρξε αυτό το θέμα των Ηνωμένων Εθνών. Θα περάσουν τρεις μήνες, θα δούμε τι γίνεται τον Αύγουστο και το θέμα είναι η κατανομή των πόρων και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ Βορείου και Νοτίου Σουδάν. Εν τω μεταξύ όμως όντως πρέπει να στέλνουμε ε, βοήθεια διότι μας μιλάτε για τον ε, Μπλε Νίλο και Νότιο Κορδοβάν μας μιλάτε ε, για τις ανθρωπιστικές δράσεις αλλά όχι ε, για την πρόσβαση της βοηθείας όπου υπάρχει τεράστια διαφθόρα και προβλήματα πρόσβασης γιατί δεν υπάρχει υποδομή και στην εποχή των βροχοπτώσεων εκτός εάν χρησιμοποιήσετε ελικόπτερα δεν μπορείτε να στείλετε βοήθεια και ε, ξέρουμε όμως ότι σε ορισμένες περιοχές θα χρησιμοποιηθεί βοήθεια ενώ σε άλλες υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και στα θέματα αυτά της προσβάσεως και της χρησιμοποίησεως θα ήθελα βοήθεια αλλά βεβαίως θα σας στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ακούσαμε θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ όμως θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα όσον αφορά την περιοχή του Σαχέλ. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στο Μαλί. Πριν από λίγο η κυρία Αλφονσίν για παράδειγμα από τους Πράσινους προσκάλεσε εδώ μία αντιπροσωπεία από τα ΜΕΝΕΛΑ την ανεξαρτησία του Σαουάτ και μας ε, μιλούσε για την δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην περιοχή όπου αντιπαλεύονται οι μουσουλμάνοι αλλά κοσμικοί με άλλες ομάδες που είναι πιο φανατικές. Υπάρχει κίνδυνος γενικότερης αποσταθεροποίησης όχι μόνο της χώρας αλλά και του Νίγηρα. Εγώ ηγήθηκα της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι εκεί που πήγαμε για τις εκλογές. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να καταλήξει να γίνει η πραγματική μποραταποθήκη. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει, τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για την περιοχή εκεί. Θέλω επίσης να επενθυμίσω ότι είναι ένα θέμα που ξεχνάμε αυτό, η Δυτική Σαχάρα δηλαδή. Εκεί θέλαμε ανθρωπιστική βοήθεια. Η χώρα μου πάνω απ' όλα, η Ισπανία. Δυστυχώς μειώθηκε πάρα πολύ. Γι' αυτό και πιστεύω ότι χρειάζεται αρρωγή αν θέλουμε να μην ξεχνιέται από τις συζητήσεις μας η χώρα αυτή. Merci. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Στίφλερ είναι η μόνιμη συγκεντριά μας για τα ανθρωπιστικά ζητήματα, γι' αυτό και της δίνω ευθύ αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θέλω να αντιδράσω, αν και όλο άκουσε είναι αλήθεια. Πράγματι, πριν από λίγο καιρό ήμουνα στο Σαέλ, στο Τσάντ πιο συγκεκριμένα. Εκεί είδα φρικτά πράγματα ε, για όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών που δεν διατρέφονται καθόλου καλά. Τα παιδιά, ε, και δεν, ούτε τα μωρά, γιατί ούτε οι μητέρες δεν τρέφονται καλά εκεί. Αλλά θέλω εδώ να υπογραμμίσω ένα πιο πολιτικό ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι σήμερα, όταν μιλάω με Ευρωπαίους πολίτες για την ε, θέρμανση του κλίματος, για τις επιπτώσεις που έχουν οι κλιματικές αλλαγές στις υπονάπτυξη χώρες, ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι με περνάνε λιγάκι, πώς να σας το πω, ε, κεντρική. Οι πολίτες των χωρών μας δεν αντιλαμβάνονται πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση αυτή. Και είμαι πεπισμένη όλο και περισσότερο γι' αυτό. Πριν μιλούσαμε για το 0,7%. Φυσικά, μπορεί να υπάρχει κρίση στην Ευρώπη, αλλά είναι σκανδαλώδε να μην έχουμε φτάσει στο 0,7%. Συχνά τη χρησιμοποιούμε άλλοθη. Μιλήσαμε για τη Γερμανία πριν, αλλά υπάρχει και η Γαλλία. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δεν είμαστε αρκετά, εντάξει ο όρος επιθετική μπορεί να μην είναι σωστός, αλλά αν μη τι άλλο να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο την αυτό που πονάει και να καταδείξουμε κάποιες αλήθειες, κάποιες πραγματικότητες που δεν μπορεί να συνεχίζουμε να γνώμε. Όσον αφορά τώρα το θάρρος των πολιτικών, εντάξει, πράγματι μπορεί να λείπει το πολιτικό θάρρος, δυστυχώς. Γιατί επιπλέον έγινε και μία δημοσκόπηση, χθε η κυρία Γιώργεβα μίλησε για αυτήν, μία δημοσκόπηση λοιπόν που δείχνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για τους πολίτες είναι μια έννοια που την εκτιμούν ιδιαίτερα και που τη γνωρίζουν όλο και περισσότερο. 90% των Ευρωπαίων πολιτών σήμερα, σε αντίθεση με 70% πριν από μερικά χρόνια, είναι υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας. Άρα οι πολιτικοί πρέπει να βρουν το θάρρος και να πάρουν τα μέτρα που πρέπει. Ο κύριος Πίβαλς, η κυρία Γιώργεβα, Ευρωπαίοι Επίτροποι που συνεργάζονται, ίσως θα έπρεπε περισσότερο ή να ε, βάλουν στο παιχνίδι και άλλους επιτρόπους και αυτό που ασχολείται με τη γεωργία, τα οικονομικά ή με άλλα θέματα, να τους βάλουν και αυτούς στο παιχνίδι. Γιατί αν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και τη θέρμανση του πλανήτη, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να δώσουμε περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα χρήματα, αλλά η κλιματική αλλαγή δεν θα αντιμετωπιστεί. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα ακόμα, αλλά θα πρέπει και εμείς, η Επιτροπή Ανάπτυξης, από την πλευρά μας, να είμαστε πιο διεκδυτικοί, να αναλαμβάνουμε και εμείς πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει να μένουμε πάντα οι τελευταίοι ή λιγότερο σημαντικοί, γιατί επειδή η Αφρική είναι μακριά, τις κλιματικές αλλαγές δεν τις νιώθουμε ακόμα εμείς στο πετσί μας πολύ. Ε, όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Ντεκάιζερ. Ότι πριν δώσουμε περισσότερα χρήματα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και ίσως να ζητήσουμε περισσότερες προϋποθέσεις, παρόλο που ο όρος προϋποθέσεις δεν μας αρέσει και πολύ. Γιατί τη χθεσινή συνάντηση, ναι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μίλησαμε πολύ για την αντοχή αυτή, την αντίσταση στις κλιματικές αλλαγές. Τώρα κατάλαβα τι σημαίνει, στην αρχή δεν το καταλάβαινα γιατί ο, όρο ο όρος αυτός στα γαλλικά resilience πολλές φορές ε, σημαίνει άλλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ σημαίνει αντίσταση, αντοχή. Πιστεύω πως τώρα πια πρέπει να μπούμε στην πρώτη γραμμή και να επιμείνουμε ως Επιτροπή Ανάπτυξης για αυτά που θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε. Η κυρία Θεοχάρους, τελευταία ερώτηση. Και μετά θα ζητήσω από τους δύο προσκεκλημένους μας να απαντήσουν συνολικά. Έχω μια γενική ερώτηση, λέει η κυρία Θεοχάρους. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την δημιουργία μιας ανθρωπιστικής task force για να μπορέσουμε να αντιδρούμε ε, πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά όταν ξεσπάει μια κρίση. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μοιράσετε τις απαντήσεις. Θα προτείνω να ξεκινήσει ο κύριος Σόρενσον, αν δεν διαφωνείτε. Κοιτάξτε, κανονικά βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο, αν και πολλές φορές ασκούμε κριτική ο ένας τον άλλο, γιατί αυτό είναι τμήμα ενός ισχυρού διαλόγου ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα ανθρωπιστικά. Για την κυρία Ντοκεζέρ και για την κυρία Στίφλερ. Εγώ δεν θα ζητήσω περισσότερα χρήματα ή δεν θα ζητούσα περισσότερα χρήματα αν δεν ήξερα ότι μπορούν να δαπανηθούν, μπορούν να χρησιμεύσουν. Έχουμε ήδη, επαναλαμβάνω, έχουμε ήδη δώσει 20 εκατομμύρια στη Συρία. Τα χρήματα αυτά με τις ροές οι οποίες υπάρχουν τώρα θα μας καλύψουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Κάποιες από τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει φτάνουν μέχρι τον Οκτώβριο, κάποιες σταματούν τέλος Αυγούστου. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη ροή της βοήθειας προς τη Συρία, καλό θα είναι να έχω λίγο περισσότερα χρήματα στη διάθεσή μου. Αν το θέμα της πρόσβασης ε, γίνει περισσότερο περίπλοκο, κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρξει σαν πρόβλημα, τότε τα χρήματα φυσικά θα διαρκέσουν περισσότερο και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να επανέλθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσω επιπλέον χρήματα πριν από το τέλος του χρόνου. Νομίζω ότι με τα χρήματα με τα οποία ζητάμε τώρα θα καλύψουμε όλες τις πιθανές δυνατότητες. Και είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στην χώρα αυτή, στη Συρία. Παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά να μην υπάρξει, θα έλεγα, περίπτωση όπου τα χρήματα της βοήθειας να χρησιμοποιηθούν για άλλους στόχους και λόγους. Αυτό θα το καλύψουμε και στα πλαίσια της εφαρμογής της αρχής της ευαισιμότητας. Για το ΣΑΚ. Το ΣΑΚ λειτουργεί πλέον τώρα, χρειάστηκε χρόνο για να λειτουργήσει και γι' αυτό το ICSC με διαβεβαιεί τώρα ότι έχουν συστήματα ελέγχου επιτόπου, που τους επιτρέπουν τα πράγματα να πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε και όχι σε άλλους. Πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια λοιπόν την οποία δίδει το Mercy Aid, η Action Contre la Faim. Ε, έχουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, έχουν δοθεί από τις κυβερνήσεις τους περισσότερο. Τώρα για τον Νότιο Σουδάν, φεύγω από τη Συρία. Το συνολικό ποσό για το 12 δεν ανταποκρίνεται στο, συνολικό ποσό το οποίο δαπανίσαμε το 11. Γιατί εμείς πιστέψαμε ότι τη στιγμή που κάναμε τον προγραμματισμό ότι η κατάσταση κάπως θα μπορούσε να βελτιωθεί. Αυτό το οποίο κάνουμε στην ουσία είναι να επανέλθουμε δηλαδή σε αυτά τα οποία είχαμε πει πέρυσι. Ο λόγος είναι ότι η κατάσταση χειροτερεύει δυστυχώς. Οι ροές δεν είναι πλήρως λειτουργικές. Πιστεύω ότι μπορούμε σε κάποιους τομείς να δραστηριοποιηθούμε καλύτερα με καταφύγια στον τομέα της υγιεινής, να βοηθήσουμε ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίες χρησιμοποίησαν τις πιστώσεις που είχαν στη διάθεσή τους για να πάρουν θέσεις σε στρατηγικά σημεία. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας σε επίπεδο λεπτομεριών. Για την κυρία Θεοχάρους, για την Task Force, υπάρχουν ε, διαφορετικές προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει. Εγώ δημιούργησα στο εσωτερικό της ΕΚΟ ένα ειδικό μηχανισμό, ο οποίος να αναζητεί τι γίνεται όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη κρίση. IT, πλημμύρες του Πακιστάν, κάτι απρόβλεπτο. Μπορώ να φέρω σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές διευθύνσεις. Είναι μια υπηρεσία η οποία είναι ήδη λειτουργική. Όπως γνωρίζετε επίσης, αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο Έχουμε και τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Αυτό συνδέεται με την ανθρωπιστική βοήθεια και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ικανότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας να συνεργάζεται στο μέλλον καλύτερα. Χρησιμοποιήσαμε τις υπηρεσίες αυτές στο σεισμό στην Τουρκία και στην αποχώρηση των πολιτών των ξένων από τη Λιβύη και αρκετοί από αυτούς είναι φυσικά δραστήριοι και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καταπολέμηση πυρκαγιών στην Ελλάδα κτλ. Οι συνάδελφοι του EEAS εξετάζουν και αυτοί με τη σειρά τους διάφορες υπηρεσίε. Έχουν μια ανθρωπιστική εντολή, αλλά από την άλλη θέλουν οι διπλωμάτες οι οποίοι είναι στη διάθεσή τους να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρα στις ε, προσπάθειές τους. Γιατί ξέρετε ότι ο πολιτικός παράγων δεν μπορεί να αγνοηθεί. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι εγώ υπεύθυνο γι' αυτά. Πάντως εδώ σας δείχνω ότι υπάρχουν τρεις ας πούμε μονάδες έρευνας χρήσιμες. Θα επανέλθουμε σε αυτά και στα πλαίσια της ρήτρα αλληλεγγύης, η οποία ζυμώνεται κάπου στα θεσμικά όργανα, Έχουμε να κάνουμε με έναν τρόπο δηλαδή εκκίνησης μιας συγκεκριμένης προσπάθειας και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ένωσης. Ο Τζόρτζ. Ευχαριστώ Κλάς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Το θέμα το οποίο υπογραμμίστηκε είναι το θέμα της πρόσβασης. Το θέμα της πρόσβασης είναι καθοριστικό να πω ότι στις καταστάσεις τις οποίες παρουσίασε ο κύριος Σέρενσεν, για την Αφρική δηλαδή, η φυσική πρόσβαση είναι πάντα κάτι το πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα η πρόσβαση στο Βόρειο Μαλί πάρα πολύ δύσκολη, στο σύνολο της κεντρικής και νότιας Σομαλίας, στον Ήγυρα Έχουμε με τη μεσαία περιοχή του Βορρά, Τάουα, στην οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση λόγω των προβλημάτων ασφαλείας στην περιοχή. Αλλά πρόεδρε, αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω τρεις τρόπους και τρεις δυνατότητες πρόσβασης. Ο πρώτος είναι η λεγόμενη λειτουργική πρόσβαση, όπου τα θέματα ασφαλείας δεν είναι το εμπόδιο. Σε αυτή τη φάση στον Άνω Ήλο και στο κράτος ε, Unity και σε άλλες περιοχές στην Μπουρκίνα Φάσο δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση λόγω των λειτουργικών συνθήκων, δηλαδή την καταστροφή των δρόμων από τις βροχές. Αυτός είναι ο ένας τρόπος πρόσβασης. Ο άλλος είναι ε, η πρόσβαση σε υπηρεσίες που σώζουν ζωές. Σε όλες τις καταστάσεις που παρουσίασε ο κύριος Σόρενσεν και εγώ υπάρχουν τρία θέματα. Το πρώτο είναι τα τρόφιμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς έχουμε πρωτοποθετήσει προσότητες τροφίμων δεξιά και αριστερά. Αλλά βέβαια επί τη βάση των στοιχείων τα οποία δυστυχώς έχουν διπλασιαστεί από πέρυσι. Δεύτερον, πρόσβαση σε νερό. Ιδιαίτερα στην Πορκίνα Φάσο, στον Ήγυρα. Εμείς ε, εδώ καλύπτουμε ένα κόστος το οποίο φτάνει περίπου 5.000 ε, δολάρια ανά ταξίδι των βιτίων, των βιτιοφόρων, πάρα πολύ ακριβό. Και τέλος χρειάζεται και υψηλότερη και δυνατότερη πρόσβαση σε πόρους, σε χρήματα και γι' αυτό εδώ απαντώ ε, την δική σας ερώτηση. για τους πρόσφυγες στο Μαλί και για τις τέσσερις χώρες στις οποίες αναφέρθηκα ήδη, Μαυριτανία, Νίγηρα, Μπουρκίνα, Φάσο και Αλγερία, Αφήνοντας την Αλγερία, γιατί εκεί η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της, οι απαιτήσει οι οποίες υπάρχουν είναι 150 εκατομμύρια δολάρια από τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου χρειαζόμαστε κατεπηγόντως 50 εκατομμύρια δολάρια. Αν δεν δώσουμε τα χρήματα αυτά, τότε θα ξεμείνουμε στις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η τελική ημερομηνία, από όπου και μετά δεν θα έχουμε χρήματα. Οι κάτοικοι, για τους κατοίκους του Νοτίου Σουάν απαιτούνται 165 εκατομμύρια δολάρια. Εμείς έχουμε στη διάθεσή μας 16 εκατομμύρια. Από τώρα λοιπόν και μέχρι την κρίσιμη περίοδο των βροχών χρειαζόμαστε 48 εκατομμύρια ακριβώς για τη λειτουργική πρόσβαση. Πετάμε τα προϊόντα εκεί γιατί δεν μπορούμε να τα πάμε οδικός. Και θα κλείσω με αυτό να πω ότι χρειάζεται κάθε βοήθεια και μέσω της κυρίας Σόρενσεν, του κυρίου Σόρενσον συγγνώμη, και μέσω των κρατών μελών να βελτιώσουμε όλες αυτές τις μορφές πρόσβασης. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ξέρω είναι ασφαλισμένοι για αυτά που κάνουν, ούτε εμείς εξάλλου, οι δύο κύριοι. Εν περιπτώσει για όσους αρχίζουν και δείχνουν τα πρώτα σημάδια εξάντλησης, να ξέρετε ότι έχετε τρεις ώρες στη διάθεσή σας, να πάρετε τις δυνάμεις σας και να επιστρέψετε στις τρεις ακριβώς, ώστε με νέες δυνάμεις να συνεχίσουμε. Έληξη η συζήτηση και καλή σας όρεξη.